Ε, συνεργασία και περνάμε στην εξήγηση ψήφων. Για την έκθεση Μπουσουτήλ σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ Μπαρμπάντος ζήτησε Εξήγηση ψήφου ο κύριος Ιντάλγκο. Πρόεδρε, δεν κατάλαβα καλά, αναφερθήκατε σε μένα. Αναφέρεστε, αναφερθήκατε σε μένα για την εξήγηση ψήφου. Ναι, ναι, έχετε ένα λεπτό για την έκθεση Μπουσουτήλ, εξήγηση ψήφου. Ναι, Πρόεδρε, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ψήφισα υπέρ για όλες τις άλλες. Γιατί θεωρώ ότι είναι καλό να, υπε... να ξεπερ... διακόπτεται ο μιλητής. Παρακαλώ, παρακαλώ, αποχωρήσατε ησύχω διότι δεν μπορούμε να ακούσουμε τον ομιλώντα. Sí. Sí, sí la superación de υπέρ όλων των λοιπόν εκθέσεων, διότι είναι σωστό να υπάρξει απελευθέρωση και άρση των ε, διατυπώσεων. Για όλες αυτές τις χώρες λοιπόν δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις καλές σχέσεις που έχουμε με αυτές τις χώρες για όλες αυτές τις ε, φιλικές, επαναλαμβάνω, και κυρίαρχες χώρες ε, την συμφωνία αυτή. Αλλά με την πανδημία στο G20 συζητήθηκε το θέμα αυτό και έτσι με αυτές τις ενεργείες συνεισφέρουμε στην οικονομική κρίση. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να πλήξουμε, να καταπολεμήσουμε ας πούμε τους φορολογικούς παραδείσους. Κάναμε, αλλά ας μην ε, απατώμεθα. Υπάρχει περίπτωση Γκούρτελ που αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους φορολογικούς παραδείσους. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία που έχουμε εδώ εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίδεται για μια πιο ευρεία και συμπεριληπτική και αποτελεσματική πολιτική κατά των φορολογικών παραδόσεων. Ευχαριστώ κύριε Μάσεπ για τη δήλωσή σας. Περνάμε τώρα στην εξήγηση ψήφου του κυρίου Σικέρσκη Άνταμ για την έκθεση Κοέλιο σχετικά με τον μηχανισμό αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου Σέγγεν. Κύριε Πρόεδρε, το καθεστώς Σέγγεν ε, είναι ποιοτικά ιδιαίτερα σημαντικό και καλό για τα κράτη-μέλη παρότι έχει τεθεί σε ισχύ μόλις πρόσφατα. Μερικές φορές ε, ξεχνάμε ότι η ελεύθερη μετακίνηση είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι ένα περαιτέρω επίτευγμα της ε, ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους, γιατί υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Υπάρχουν πολύ υψηλοί περιορισμοί όσον αφορά τις ε, όμορες χώρες. Αυτό αφορά κυρίως την Πολωνία και την Λετονία. Υπάρχουν περιορισμοί στη μετακίνηση και προς Ανατολά, στην Ανατολική πλευρά, κυρίως με χώρες με τις οποίες έχουμε ιστορικούς ε, πολιτικούς ε, δεσμούς, δεσμούς γειτονίας. Παράλληλα, ε, με το Σέγγεν εισήχθηκε ένα κοινό σύστημα ελέγχου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το σύστημα ελέγχου την χάνει υπερβολικής εκμετάλλευσης και αυτό δεν βοηθά στο να προβληθεί μια θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Finito. Ευχαριστώ τον κύριο Σικέρσκι. Δεν ζητούν άλλοι συνάδελφοι εξήγηση ψήφου, οπότε διακόπτουμε. Καλή όρεξη σε όλους.